Hello. It's half past uh, Καλησπέρα. Είναι τρισήμιση, αλλά υπάρχουν εδώ στην αίθουσα ήδη κάποιοι συνάδελφοι. Λίγοι, ελάχιστοι. Τρεις, τέσσερις. Τέσσερις τουλάχιστον. Θα περάσω στα πορτογαλικά. Είμαστε λίγοι βουλευτές ακόμα εδώ. Δεν έχουν έρθει αρκετοί. Αφήσαμε και λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσουμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Έχει διερμηνία. Εντάξει. να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, ελπίζοντας ότι μεταξύ θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. Ως προς την ημερήσια διάταξη και αυτά που προβλέπει, σημείο πρώτο η έγκριση αυτής, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις την εγκρίνουμε και περνάμε στο σημείο 2 έγκριση των πρακτικών της 24ης Μαΐου. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ή διαφωνίες να τις επισημάνετε. Εφόσον δεν φαίνεται να υπάρχουν, τα εγκρίνουμε. Δεν έχω ανακοινώσει ως πρόεδρος. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο σημείο προσυζήτηση έκθεση της Επιτροπής Γυναικών με ποιου τρόπου μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ήπεθρο. Η συγγήτρια κυρία Κέστιγκελ. Θα έχουμε μια πρώτη συζήτηση περί των τροπολογιών της έκθεσης. Ο λόγος στην εισηγήτρια για να κάνει τις απαραίτητες παρατηρήσεις ως προς τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε. Ήδη έχει γίνει μία πρώτη συζήτηση επί του περιεχομένου της έκθεσής μου. Συζητήσαμε δηλαδή την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, η οποία ασχολείται με την ισότητα των και την κοινή αγροτική πολιτική. 75 τροπολογίες υπέβαλαν οι συνάδελφοι, οι οποίες τροπολογίες θεωρώ πως αφορούν αρμοδιότητες που δεν είναι αυτής της Επιτροπής. Έχουμε ξεπεράσει δηλαδή την ε, δική μας αρμοδιότητα και νομίζω πως έχουμε χάσει την ε, εστίαση στο θέμα μας. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες πολιτικές απόψεις που φαίνονται σε αυτές τις τροπολογίες. Ε, σε όσο επιτοπλίστων ασχολούνται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο χώρο της γεωργίας, εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργία δικτύων, δημιουργία των ε, αναγκαίων υποδομών έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να συνδυάσουν την ε, οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, κάτι που και εμείς συζητάμε στη γνωμοδότηση. Αναφέρονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία καταφέραμε να συμπεριλάβουμε με μορφή συμβιβασμού σε δέκα συμβιβαστικές τροπολογίες. Τονίζεται επίση ο πολύ σημαντικό ρόλο των γυναικών στην ε, Ήπεθρο. Υπάρχουν όμω κάποιε τροπολογίε τι οποίε δυστυχώ δεν μπόρεσα να ε, αποδεκτώ από ορισμένου και όδες συζητητέ οι οποίοι προέρχονται από άλλε πολιτικέ κατευθύνσει, άλλου πολιτικού χώρου από εμένα, ορισμένε που αναφέρονται στην επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα. Σε γενικέ γραμμέ, οι γυναίκε πρέπει να θεωρούνται ως επιχειρηματίες όταν δίκουν μια γεωργική εκμετάλλευση, όταν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις για την επιχείρησή τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες τις οποίες θα ήθελα να σχολιάσω. Υπάρχουν ορισμένες που αναφέρονται σε ειδικά προγράμματα για τις γυναίκες στην Ήπεθρο στα πλαίσια του ε, Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχουν λοιπόν κάτι τέτοιο, κάτι... κάποιες τροπολογίες οι οποίες ζητούν δυνατότητες οι οποίες ήδη προβλέπονται από τα διάφορα ταμεία. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες για πρόθεση των γυναικών. Υπάρχει ο κανονισμός 1305 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την στήριξη της υπαίθρου μέσω των ταμείων. Και ε, αυτό το ξέρω πολύ καλά, διότι και εγώ υπήρξα μέλος της ε, ομάδας που ασχολήθηκε με αυτές τις δυνατότητες και επί δύο χρόνια διαπραγματευόμασταν αυτές τις ε, συγκεκριμένες δυνατότητες στήριξης των γυναικών στην Ήπεθρο. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι αυτές οι τροπολογίες ίσως είναι κάπως περιτές εδώ επειδή ήδη προβλέπονται παρόμοια μέτρα. Το θέμα είναι να δούμε πού μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πού υπάρχει λοιπόν περιθώριο βελτίωσης, πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, κονδύλια από τα μία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην ε, κοινοτική πολιτική. Υπάρχουν τροπολογίες σχετικές με αυτό, ωστόσο δεν θεωρώ πως θα μας οδηγήσουν στο στόχο που θέλουμε. Η αγροτική πολιτική, οι τιμές ε, των γεωργικών προϊόντων αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε περίοδο κρίσης και χρειάζεται να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Όμως πιστεύω πως η συνεκτίμηση της διάστασης του φίλου ίσως δεν είναι τόσο σχετική με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι γυναίκες εδώ έχουν άλλα προβλήματα από ε, αυτό το gender mainstreaming. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως ε, πρέπει να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη. Υπάρχουν βέβαια πολλές ε, επικοδομητικές προτάσεις για κατάρτιση, για ισχυρότερη δικτύωση των γυναικών στην ύπεθρο, για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, Πιστεύω λοιπόν πως αυτές τις τροπολογίες πρέπει να τις στηρίξουμε και η γνωμοδότησή μας θα βοηθήσει την αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Γεωργία. Ελπίζω και ελπίζω ορισμένα σημεία που αναφέρονται στην γνωμοδότησή μας να συμπεριληφθούν στην στο τελικό σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Γεωργία, έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση των γυναικών στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. και τις εξηγήσει για το περιεχόμενο του εγγράφου. Δεν έχουμε εδώ σκιώδει εισηγητές. Όμως ξέρουμε ότι ενημερωθήκαμε ότι ζητήθηκε από σκιώδη εισηγητή να διαβαστεί η παρέμβασή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κόστινγκερ για την προσπάθεια που κατέβαλε και τη δουλειά που έκανε, ιδιαίτερα στην προσπάθεια έβρεση συμβαστικών λύσεων και η ομάδα μας, οι σοσιαλιστές, θα ήθελε να τονίσει ορισμένα σημεία στην γνωμοδότηση. Οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής και για την δική μας ομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ε, ληφθεί υπόψη η ισορροπία και ίσες ευκαιρίες ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, ιδιαίτερα σε τομείς όπου οι γυναίκες έχουν διπλό έργο επαγγελματικό και οικογενειακό. Έχ, πρέπει να είναι στην, ε, στο σπίτι τους ταυτόχρονα και στην δουλειά. Χρειάζονται λοιπόν οι αναγκαίες υποδομές και κοινωνικές υποδομές και ψηφιακές υποδομές. Για παράδειγμα ευρυζωνικό ίντερνετ, ε, δίκτυο συγκοινωνιών και Επίσης, ε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η φυγή των ανθρώπων από την Ήπεθρο, είναι η αστικοποίηση. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθούν οι σωστές προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορεί μια γυναίκα να γυρίσει στην Ήπεθρο, να ζήσει στην Ήπεθρο και να εργαστεί εκεί. Χρειάζεται λοιπόν, ε, όπως είπα και πριν, κοινωνικές ε, υπηρεσίες συγκοινωνίες ευρυζωνικότητα, ψηφιακή σύνδεση. Για τους ε, σοσιαλιστές επίσης η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως στην κοινή αγροτική πολιτική. Θεωρούμε όμως πως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής, γι' αυτό και οι σοσιαλιστές ζητούν βελτίωση στον τομέα αυτό. Τώρα, αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι οι, τα περιοριστικές ε, είναι οι περιορισμοί στις ε, γυναίκες, ιδιαίτερα στις εργαζόμενες μητέρες. Χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Ευχαριστούμε. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι εδώ οι υπόλοιποι και εισηγητές. Η κυρία Σόντροβα νομίζω έχει ζητήσει το λόγο γιατί θέλει να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να στηρίξω την ε, γνωμοδότηση της συναδέλφου. Η κοινή γεωργική πολιτική στις ε, ζώνες της Πέθρου αναμφίβολα βοηθάει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και η γνωμοδότηση αυτή είναι, ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση, εξού και εγώ την υποστηρίζω. Όπως θα υποστηρίξω και τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι αυτές οι θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσω του κοινού ταμείου για την γεωργική πολιτική και θα πρέπει να αναπτυχθούν υπηρεσίες προς τη χρησιμοποίηση των θέσεων αυτών. Θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες δηλαδή υπηρεσίες υποστηρικτικές εις, της, εις την Ήπεθρο. και άλλες υπηρεσίες που θα βοηθούν στην απορρόφηση αυτών των θέσεων και στην καλύτερη οργάνωση της ζωής στην Ήπεθρο. Και η έκθεση καλώς έχει, αλλά είναι σωστό να μας κατανοούν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο οι πολίτες. Το γεγονό δηλαδή ότι δίνουμε μια έμφαση στην ισορροπία μεταξύ τη επαγγελματική και τη ιδιωτική ζωή θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα γίνεται κατανοητό. Και αυτό προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλύτερες υπηρεσίες στις γυναίκες σε αυτές τις ζώνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πετήρ τώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Κάστιγκερ για αυτή την έκθεση Καλύπτουν τα βασικά σημεία που ε, πρέπει να καλύπτονται από ένα τέτοιο, μια τέτοιο θέμα και είναι αρκετά ισορροπή. Εδώ πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε χειροπιαστές λύσεις για τις θέσεις εργασίας στην περιοχή της Υπέθρου. Θέλουμε η Υπέθρο να είναι ένα μέρος που μπορούν να κατοικήσουν οι πολίτες, όχι να την εγκαταλείπουν μόνο. Οπότε πρέπει να υπάρχουν ε, κοινωνικά, ε, κοινωνικές ε, δομές που να ενθαρρύνουν τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να παράγουν, να παράγουν τρόφιμα, να προφυλάσσουν το περιβάλλον, αλλά από την άλλη να, ε, προστατεύουν και τις αξίες που εκπροσωπούμε. Βάσει της κοινή γεωργικής πολιτικής υπάρχουν μέσα και εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και θα πρέπει και τις καινοτόμες ε, ιδέες να τις καλλιεργήσουμε περαιτέρω, όπως την προσφορά υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση ώστε όσοι κατοικούν στην Ήπεθρο ε, και παράγουν τρόφιμα να μπορούν να έχουν κατανάλωση και σε αυτό το επίπεδο, στην Ήπεθρο και να προσφέρουν και υπηρεσίες όπως ε, τουρισμό στην Ήπεθρο, αγροτουρισμό και άλλε κοινωνικέ υπηρεσίε, λόγω χάρη οίκους ευγυρία ή νηπιαγωγία και βρεφονιπιακούς σταθμού για τα παιδιά. Ε, η εντύπωση μου είναι ότι υπάρχει ευρύ πεδίο για να αξιοποιήσουμε τα υπάρχοντα μέτρα και να τα υλοποιήσουμε και υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε περαιτέρω θέσει εργασία στην Ήπεθρο για τι γυναίκε. Αυτό για μα είναι ήδη σημαντικό όπως και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και ε, το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι κατοικούν, η αιστεία τους βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, οπότε έτσι διαφυλάσσουν τις περιοχές αυτές ως κάτοικοι. Ως προς την κυρία Κέστιγκερ λοιπόν θα την υποστηρίξω στην έκθεση αυτή διότι πιστεύω ότι μπορεί να διευκολύνει τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο και να τους προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και καλύτερες δουλειές. Επίσης θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και άλλα σχετικά θέματα. Μόνο 20% των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη είναι εκμεταλλεύσεις που χειρίζονται γυναίκες και είναι πολύ μικρό ο αριθμό όσων εργάζονται όντω στον τομέα τη γεωργία. Ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη πιο πολλή δουλειά λοιπόν προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Ο λόγο στην κυρία Μέρκελ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Κιώστινγκερ για την γνωμοδότηση. Έχει συμπεριλάβει αρκετά στοιχεία τα οποία είχαμε ζητήσει. Ωστόσο, με ανησυχεί το ότι όπω είπε και προηγουμένω, υπάρχουν υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θεωρεί υπερβολικά και τα οποία αφορούν την ισότητα των φύλων. Όμως εδώ είμαστε σε μια επιτροπή η οποία ακριβώς με αυτό ασχολείται, με την ισότητα των φύλων. Η Επιτροπή Γυναικών δεν είναι μια ε, υποεπιτροπή της Επιτροπής Γεωργίας, ούτε υποεπιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα, για την απασχόληση. Είναι μια συγκεκριμένη επιτροπή που έχει ε, ως κεντρικό άξονα την ισότητα των φύλων. Και εδώ ασχολούμαστε με τις γυναίκες οι οποίες εργάζονται στον τομέα της γεωργίας. Όμως υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες ε, μπορεί να μην είναι αγρότες, ζουν όμως στην Ήπεθρο. Και αυτές βρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση με τις ε, αγρότες χωρίς να εργάζονται σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό λοιπόν ε, σίγουρα μπορώ να πω ότι πράγματι υπάρχει κρίση στην Γεωργία. Όλοι μας γνωρίζουμε το θέμα με τις χαμηλές τιμές του γάλακτος. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές ε, διαστάσεις, πολλές ε, πτυχές, όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση έχει μια διαφορετική διάσταση στην Ελλάδα, ας πούμε, από ό,τι στη Γερμανία. Υπάρχει Υπάρχουν και διαφορετικές διαστάσεις στην αγροτική πολιτική. Πρέπει λοιπόν ε, επομένω, να καταστεί σαφές ότι όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για μια γεωργική εκμετάλλευση, όσο πιο δύσκολα τα, βγάζει, τα βγάζουν πέρα οι αγρότες, τόσο πιο δύσκολη είναι η θέση των γυναικών εκεί. Επίσης, ε, η ισότητα πρέπει να υπάρχει παντού. Όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν προβλήματα στον ε, χώρο της ε, γεωργίας. Προβλήματα τα οποία δεν αφορούν μόνο οικονομικούς παράγοντες αλλά και την ε, ενδοοικογενειακή βία για παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται στήριξη σε όλες ανεξάρτητως τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποια από τις υπόλοιπες συναδέλφους να κάνει κάποιο σχόλιο για την έκθεση. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε σε πολλά θέματα. Η συνάδελφος από τους σοσιαλιστές έχω να πω ότι δεν ήταν παρούσα κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και γι' αυτό λοιπόν ίσως δεν μπορεί να έχει και προσωπική άποψη. Σίγουρα τις μεταφέρθηκαν ε, οι πληροφορίες από τους βοηθούς της, όμως να, να πω και εδώ ότι η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή έχει ήδη συζητηθεί. Αναφέρθηκε ε, ο, δυσανα, το, ο δυσανάλογος φόρτος εργασίας σε γυναίκες οι οποίες ε, εργάζονται σε μια ε, γεωργική εκμετάλλευση και πρέπει πρέπει να συνδυάσουν οικογένεια, προσωπική ζωή και ε, δουλειά. Θεωρώ λοιπόν πως είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θεωρώ επίσης πως είναι ε, αυτονόητο ότι οι γυναίκες συνεισφέρουν πάρα πολύ σημαντικά στην γεωργία. Δεν χρειάζεται λοιπόν επιπλέον αναφορά τώρα. Εμείς κάνουμε μία γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά μία έκθεση η οποία έχει ως τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ήπεθρο, σε αγροτικές περιοχές». Και ίσως είμαι αφελής, αλλά θεωρώ πως η γνωμοδότησή μα πρέπει να ασχοληθεί ακριβώς με το πώς μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στην Ήπεθρο. Φυσικά και θα σταθούμε στις γυναίκε. Φυσικά και συνεπάγεται ότι πρέπει να βελτιωθεί η θέση των γυναικών, όμως πιστεύω πως δεν είναι ανάγκη να ξεφεύγουμε από την ουσία. Τώρα, φυσικά και υπάρχουν διαφορές ε, στα κράτη-μέλη και για ιστορικούς λόγους και για άλλους. Το αν οι γυναίκες έχουν στην κατοχή τους ε, γη, αυτό οφείλεται σε πολλούς ε, λόγους ιστορικούς, για παράδειγμα στην περίπτωση της Ανατολικής Ευρώπης. Σε άλλα κράτη-μέλη, οι γυναίκες ιδιοκτήτε γεωργικών εκμεταλλεύσεων ε, δεν είναι 28% αλλά ξεπερνά το 50%. Αυτό έχει να κάνει με διάφορους λοιπόν λόγους όπως σας είπα, με τι διάφορες υποδομέ που υπάρχουν. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα πιστεύω πως έχουν διαφορές και ως τέτοια θα μας κάνουν να χάσουμε την ουσία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναλωνόμαστε στο πόσο επί της 100 ποσοστό ιδιοκτησίας έχουν οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να πω πως ε, είχαμε μια καλή συνεργασία με τις άλλες πολιτικές ομάδες, με τους σκιώδεις ηγητές και υπήρχε θέληση από ό,τι είδα να δουλέψουμε την γνωμοδότηση, να δούμε πώς μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στην Ήπεθρο στον χώρο της Γεωργίας. Και αύριο θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση και ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να ψηφίσουμε θετικά και να παραδώσουμε μια ε, επικοδομητική γνωμοδότηση στην Επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω λοιπόν την ε, εισηγήτρια για την επεξεργασία των τροπολογιών που βλήθηκαν και όλου του συναδελφού είναι το λόγο για να κάνουν τι παρατηρήσει του και τη γραμματεία τη Επιτροπή ΦΑΜ που εργάστηκε για το θέμα. Προφανώς ε, οι κάποιες αποκλήσεις απόψεων που καταγράψαμε σήμερα εδώ στη συζήτηση ελπίζω ότι αύριο θα αντικατοπτριστούν και στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Μετά από το σημείο αυτό μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο της ημερήσιας διάταξης ανάγκη για στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλυφθούν οι ανισότητες της συντάξης βάσει του φύλου. Η συγγήτρια κυρία Λεγκρίπ. Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα δούμε για πρώτη φορά την έκθεση. Το κείμενο που μας υποβάλλει η κυρία Μανουέλα Σαμέκ Λοντοβίση. Δεν ξέρω αν ήθελε η κυρία Λεγκρίπ να μας ε, κάνει κάποιες πρώτες παρατηρήσει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. 38% αυτό το μέγεθος θέλω να σας δώσω. Δηλαδή 38 ευρώ για κάθε 100 ευρώ. Αυτό αποτυπώνει την ενισότητα των συνταξιών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 38%. Πρόκειται για μια τεράστια και απογοητευτική απόκληση και αυτό το είχαμε συζητήσει και με τις άλλες ομάδες, να επικεντρωθούμε δηλαδή επί της απόκλησης αυτής μέσω μιας γνωμοδότησης ε, πρωτοβουλίας που είχα την τύχη να είμαι η συγκεντριά της τελικά. Οι διάφορες πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή μας ε, νομίζω ότι για μια φορά εδώ συγκεντρώνουν απόλυτη ομοφωνία επί του μεγέθους επί του γεγονότος αυτού. Η τεράστια αυτή διαφορά, η τεράστια αυτή απόκληση. Και έχουμε όλοι και όλες τη βούληση να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Και για την απόκληση τη μισθολογική, όπως και για την συνταξιοδοτική, Gender Pension Gap, λέει στα αγγλικά η κυρία Λεγκρίπ. από το 1957 είναι κατοχυρωμένη αν θέλετε η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα θέματα αυτά και επομένως αντιπροσωπεύει αν θέλετε και απόκληση στο πλαίσιο του δικαίου. Και εδώ έχουμε έναν ε, συμπληρωματικό κίνδυνο που βαραίνει τις γυναίκες σε σχέση με την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν έναντι τις οποίες είναι ακόμα πιο εκτεθειμένες. Έχουμε την προσωπική τους κατάσταση, την οικογενειακή τους κατάσταση, μπορεί να είναι διαζευμένες, παντρεμένες, χείρες, μπορεί να έχουν παιδιά, να μην έχουν κτλ. και οι ανήπαντες μητέρες στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζουν μια καταστροφική κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τον έγγραφο εργασία που επεξεργαστήκαμε με την εξαιρετική βοήθεια της ε, γραμματείας ένα πρώτο έγγραφο προκειμένου να σκιαγραφίσουμε κάποιες κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε, να αποτρέψουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν μιλούμε για κάποια καταπολέμηση ε, διαγενειακή, μιλούμε για την άμεση αντιμετώπιση τη σημερινής κατάστασης και την αποτροπή της μελλοντική κατάστασης προκειμένου να μην συνεχιστεί αυτή η απόκληση. Και θα ήθελα σχετικά με το πεδίο της μελέτης μας να πω ότι εδώ δεν συζητούμε ώστε να ανταλλάσσουμε γενικές απόψεις σχετικά με το συνταξιωτικό σύστημα, αλλά προκειμένου να επιφέρουμε συγκεκριμένες απτές προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της απόκλησης της συνταξιωτικής μεταξύ των ανδρών και των γυναικών που είναι θέμα αρμοδιότητος μάλλον η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά περιορισμένη στο θέμα εδώ εξαιρετικά περιορισμένη πρέπει να δούμε λοιπόν ποια εργαλεία μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας που να εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μας να αποτρέψουμε, επαναλαμβάνω για το μέλλον την απόκληση της συνταξιότητα αυτή, απόλυτα σεβόμενη βεβαίως την αρχή της επικουρικότητας και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις αρμοδιότητές τους. Και ήθελα να θυμίσω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις πολιτικές ομάδες. Η οργάνωση, η δομή του συνταξιωτικού συστήματος είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια επικουρική αρμοδιότητα επί τη βάση του άρθρου 153 της Συνδικής. Και βρισκόμαστε σε αυτό το στενό και πολύ συγκεκριμένο ορισμένο πλαίσιο. Γιατί λοιπόν είναι απαραίτητη η αποτροπή του φαινομένου αυτού. Το 38% που σας ανέφερα από την αρχή παραπέμπει σε πρόσφατες μελέτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε κατηγοριοποιήσει την απόκληση αυτή για τους 65 και άνω ετών. Δηλαδή την απόκληση μεταξύ των φύλων στα συνταξιωτικά θέματα. Που είναι ανεξάρτητο θέμα από, το, από τη μισθολογική όπως σας έλεγε απόκληση. Και μιλούμε για τα μεγέθη πριν από τους φόρους που λαμβάνουν οι γυναίκες σε σύγκριση με τα αντίστοιχα που λαμβάνουν οι άνδρες. Και έχουμε εδώ μια έντονη τάση εντός ε, του μεγέθους της απόκλησης αυτής να έχουμε τις πιο εκτεθειμένες κατηγορίες Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση γυναικών σε αυτές τις ομάδες 1,9 γυναίκες ανά έναν άνδρα μέχρι τρεις γυναίκες ένα έναν άνδρα. Δηλαδή έχουμε μια έντονη υπερσυγκέντρωση γυναικών έναντι των ανδρών στις χαμηλότερες εισοδηματικές συνταξιδοτικές κατηγορίες. Και θα πρέπει κανείς εδώ να ζυγίσει μετρήσιμους παράγοντες, μετρήσιμους δείκτες, προκειμένου να μπορέσει να σταθμίσει ακριβώς την απόκληση. Η απόκληση αυτή απορρέει από πάρα πολλά μειονεκτήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου γυναίκες. Και μεταξύ των μειονεκτημάτων αυτών υπάρχει και η μισθολογική απόκληση Gender Pay Gap. Ακούμε πάλι στα αγγλικά. Διότι υπάρχει άμεσος σχετισμός μεταξύ του μέσου μισθολογικού επίπεδου που λαμβάνει κανείς και του συνταξιδοτικού του επίπεδου. Ο σχετισμός όμως αυτός μεταξύ του, της μισθολογικής απόκλησης και της συνταξιωτικής απόκλησης δεν έχει αν θέλετε αποτυπωθεί με απόλυτα επιστημονικό και στατιστικό τρόπο. Διότι αφενός έχουμε δεδομένα που πάρα πολύ συχνά δεν είναι συγκρίσιμα και αφετέρου παρατηρεί κανείς εμπειρικά μια πολύ μεγάλη διαφορετικότητα, ποικιλότητα καταστάσεων. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλες αποκλήσεις μισθολογικές αλλά αντίστοιχα σχετικά μικρές συνταξιδοτικές. Και το αντίστροφο, δηλαδή υπάρχουν χώρες όπου η μισθολογική απόκριση είναι περίπου ανεκτή αλλά η συνταξιωτική καθόλου. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών αυτή τη στιγμή. Μεταξύ των 28 κρατών μελών. Αν δούμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένε Πολιτείες δηλαδή, η μείωση της μισολογικής απόκληση δεν συνοδεύεται που έχει σημειωθεί στι ΗΠΑ, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση της συνταξιωτική απόκληση. Πρόκειται λοιπόν ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό, το οποίο απαιτεί μια συνολική, σφαιρική όπως λέμε συχνά προσέγγιση προκειμένου να αντιμετωπίσει κανείς όλους αυτούς τους παράγοντες διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν λόγω των μέσων μισθολογικών τους εσόδων και τα συνταξιοδοτικά τους έσοδα. Οι διάφοροι αυτοί παράγοντες που εξηγούν την απόκληση αυτή μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες Υπάρχουν και πολλές άλλες. Μια αντελεχής μελέτη θα μας επέτρεπε περισσότερα ευρήματα. Έχουμε την συνεχιζόμενη μισθολογική απόκληση. Έχουμε μια μικρότερη διάρκεια πραγματικής εργασίας με διακοπές που οφείλονται σε διάφορους λόγους αλλά στις γυναίκες απαντώνται πιο συχνά και έχουμε μια δυσανάλογη τάση των γυναικών να εργάζονται μερικώς, με μερική απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες. Και είναι και αυτός ένας παράγων που έχει σημαντικό αντίκτυπο επί των μελλοντικών συνταξιωτικών τους εσόδων. Στο έγγραφο εργασίας που έχουμε υποβάλει Προτείνουμε κάποιε ιδέε λοιπόν και κάποιε κατευθύνσει για την διαμόρφωση τη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αποτροπή του φαινόμενου αυτού. Αλλά βεβαίω θα ήθελα να έχουμε μια ευρύτατη συζήτηση, την ευρύτερη δυνατή και απευθύνομαι και στου εκπροσώπου των άλλων πολιτικών ομάδων, όπω και στην Επιτροπή Απασχόληση βεβαίω, η οποία ασχολείται και αυτή με το θέμα και εμεί θα προσπαθήσουμε υπό το φως της μελέτης που έχει αναθέσει η Επιτροπή ε, Γυναικών που θα την παρουσιάσουμε σε λίγο. Θα έπρεπε λοιπόν, προκειμένου να επεξεργαστούμε με αποτελεσματικό τρόπο μια τέτοια στρατηγική ευρωπαϊκή για την αποτροπή του φαινομένου αυτού, πρώτον, να έχουμε αξιόπιστους δείκτες, να εντοπίσουμε αξιόπιστους δείκτες, και να έχουμε αυξημένη προσοχή για ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες διότι οι γυναίκες πάρα πολύ συχνά δεν είναι ενήμερες για με την κατάσταση αυτή. Δεν είναι απολύτως ενήμερες. Πρέπει λοιπόν να είναι προετοιμασμένες προκειμένου να έχουν αναλάβει τακτικές, στρατηγικές αντιμετώπιση του φαινόμενου αυτού. Επίσης, χρειάζεται μια εντατικοποίηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την ισότητα των φύλων. Χρειάζεται όμως η πραγματική παρακολούθηση της εφαρμογής των οδηγιών από πλευρά των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε το θέμα της ε, αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής του συνόλου της εθνικής νομοθεσίας που υφίσταται σχετικά με τα θέματα αυτά εκτός από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αλλά βεβαίω το να βρούμε δείκτες, το να προσέχουμε και να ευαισθητοποιούμε σχετικά με το ζήτημα Και εδώ μου έρχεται στο νου το φύλλο πορεία ε, σχετικά με την ισορροπία ε, ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου ε, της Επιτροπής που είναι μια στρατηγική που στοιχειοθετεί μια καλή βάση εκκίνησης σχετικά με την αντιμετώπιση και του θέματος αυτού. Χρειάζεται λοιπόν μια πραγματική υποστήριξη σχετικά με τα συνταξιωτικά συστήματα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να υπάρξει βαθμιαία μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αποτραπούν αυτά τα φαινόμενα που συνεισφέρουν στη διατήρηση της απόκλησης αυτής. Αυτά ήταν κάποια στοιχεία, συνάδελφοι, προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε μια την πλαίστερη δυνατή στρατηγική για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Για τα επόμενα βήματα να πω το εξή. Θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα επί του εγγράφου εργασία και προτείνουμε μια νέα ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου πλέον της νομοδότησης 10 και 11 Οκτωβρίου στη συνεδριάση της Επιτροπής και θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και με τους κοιόδης. Να ορίσουμε δηλαδή για μια ημερομηνία υποβολής των τροπολογιών ώστε τέλη Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου, να έχουμε άλλη μία συνειδριέση για να εξετάσουμε και τις τροπολογίες προκειμένου διατηρώντας φυσικά και το χρονοδιάγραμμα των ε, συναντήσεων του Σκιώδης Κιώδης, εν για να είμαστε έτοιμοι για τις αρχές του 17, τον Ιανουάριο του 17, θα ακούσω με μεγάλη προσοχή τις συνεισφορές των συναδέλφων εν ώψη και τις παρουσίες που θα έχουμε σε λίγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστούμε. Πρωτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να δώσω το λόγο στην κυρία Λαντοβυσή για να μας παρουσιάσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα σας παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα της μελέτης. Είναι μια σύντομη μελέτη η οποία ε, παρουσιάζει μια επισκόπηση των πρόσφατων αλλαγών στα συνδιοπιστωτικά συστήματα με από την οπτική γωνία του φύλου και τις διάφορες προβλέψεις από συγκριτικές μελέτες για το συνταξιδοτικό αυτό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο αρχικά είχε εκτιμηθεί από μία μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του οποίου εννοώ. και είδαμε ότι σωστά αντικατοπτρίστηκε ε, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η έκθεση αυτή της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής σε σχέση με τις τάσεις που επικρατούν στα συνταξιδοτικά συστήματα και τις διάφορες αποκλήσεις που υπάρχουν. Τι έλεγα, το χάσμα στις συντάξεις εκτιμήθηκε πρώτη φορά το 2013. Μια έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Justice προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα κοιτάζω την ε, γενική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και ούτω καθεξής για τις τάσεις της συντάξης που χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία ε, για να ε, αντικατοπτρίσει και τις επιπτώσεις που έχουν οι αλλαγέ στα συνταξιδοτικά στα δύο φύλλα και τη σύγκριση μεταξύ τους. Οπότε φαίνεται ότι έχουν εισακουστεί ε, οι παρατηρήσεις μας. Πρώτα απ' όλα λίγα λόγια για τις πρόσφατες συνταξιδοτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές έχουν επιταχυνθεί ιδιαιτέρως λόγω των πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων και των τάσεων γύρανσης του πληθυσμού που ασκούν πιέσεις, πιέσεις για αλλαγές στα συνταξιδοτικά συστήματα και προκειμένου να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών. Ταυτόχρονα η κρίση, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχουν δείξει ότι υπάρχουν προβλήματα από προηγούμενες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε κάπως να αντιμετωπιστούν. Τα βασικά προβλήματα που έχει δείξει η κρίση να υπάρχουν έχουν να κάνουν με ε, τους κινδύνους που προκύπτουν λόγω έλλειψης προσαρμογής οι προηγούμενες ε, εκδοχές μεταρρυθμίσεις είχαν να κάνουν με τις εισφορές περισσότερο και την προχρηματοδότηση κάποιων συστημάτων, δηλαδή το συνδυασμό ιδιωτικών με δημόσιες πηγές μετακινηθήκαμε προς συστήματα με διαφοροποιημένες πηγές, μειώνοντας τον τομέα των κρατικών συντάξεων, αλλά με την κρίση αυτού του είδους η μεταρρύθμιση, η αναθεώρηση, έδειξε ότι υπήρχαν πολλές ελλείψεις, ιδίως ως προς τη σκοπιμότητα των μέτρων το ε, γενικό εισόδημα ε, κάλυψης και επειδή πολλοί έχαναν τη δουλειά τους, δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε γενικό συστήματα προστασίας και συνέχιζαν να δίνουν τις οικονομίες τους στα ατομικά προγράμματά τους για τη συνταξιδότηση. Οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν περισσότερο με την ιδιωτική διαχείριση των προσωπικών ε, συστημάτων που χρησιμοποιεί ο καθένα είχαν κυρίω επιπτώσει στα διάφορα άτομα αυτά. Δηλαδή, σε ατομικό επίπεδο αναλαμβανόταν περισσότερο κίνδυνο. Αυτό οδηγεί κάποιε χώρε, τι υποχρεώνει να μεταρρυθμίσουν το σύστημά του και να προβλέψουν περισσότερη ρύθμιση για τα προσωπικά προγράμματα συνταξιδότηση και τα επαγγελματικά τη απασχόληση. Προκειμένου να υπάρξουν κάποιες μορφές συνταξιδοτικής κάλυψης και για τις ε, ατυπικές ασυμβατικές μορφές εργασίας, για την απασχόληση σύντομης διάρκειας, για τις συμβάσεις σύντομης διάρκειας και για να αυξηθούν τα ωφελήματα των κρατικών συντάξεων σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτή η κίνηση για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συνταξιδοτικών συστημάτων ήταν η μειονότητα. Μόνο μερικές χώρες το έκαναν αυτό, οι περισσότερες προσπάθησαν να αυξήσουν περισσότερο την βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών του συστημάτων και να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αλλαγέ στα συνταξιδοτικά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς την ισότητα των φύλων. Ε, υπάρχει δυνατότητα να επηρεαστούν ιδιαίτερα στα φύλλα στη σύγκριση που κάνουμε μεταξύ τους. Κάποια από αυτά ήδη μας τα είπε η εισηγήτρια. Τα βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει προσεκτικά να εξετάσουμε όταν βλέπουμε τις επιπτώσεις των συνταξιδοτικών συστημάτων στα δύο φύλλα είναι ο μεγαλύτερο συσχετισμός μεταξύ των διαβίου εισφορών και των εισοδημάτων από τη σύνταξη και η κίνηση προς ένα σύστημα με διαφορετικούς πυλώνες όπου συνδυάζουμε τα ιδιωτικά προγράμματα με τα προγράμματα που προκύπτουν που προσφέρουν κάλυψη λόγω τη απασχόληση κάποιου. Για να έχει κανεί καλά στα εξωτερικά ωφελήματα πρέπει να έχει δουλέψει πάρα πολύ. Να έχει πολλά χρόνια στην ενεργό απασχόληση και κατά προτίμηση στην απασχόληση πλήρου χρόνου, όχι στην μερικού χρόνου, διότι ο όγκο ωφελημάτων που αποκομίζουν οι άνθρωποι όταν φτάνουν στη σύνταξή του αντιστοιχεί κατά πολύ τις αποταμιεύσεις στις οικονομίες και τις εισφορές που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματική του σταδιοδρομίας στο εξωτερικό του ταμείο. Ε, όπως γνωρίζουμε λοιπόν, οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλότερες, ε, συντομότερες ε, σταδιοδρομίες επαγγελματικές, ε, πολλές φορές σύντομης διάρκειας και κυρίω οι γυναίκες που προσφέρουν φροντίδα. Δεν μπορούν να δουλέψουν ε, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Οπότε με αυτές τις αλλαγές, ιδίω, ε, οι γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα ή τα άτομα με διακεκομένες σταδιοδρομίες βασίζονται πολύ περισσότερο τις ελάχιστες συντάξεις και μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα φτώχεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτές οι αλλαγές είναι σημαντικές και θα επηρεάσουν πολύ και τις διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τις συντάξεις. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ενίσχυση της αρχής της αναλογιστικής ε, προσέγγισης στα συντοξιωτικά συστήματα. Ως προς τις συντάξει, ε, παίρνεις αυτό που κατέβαλες, αυτό που κατέβαλες ως εισφορά. Στην ε, τρίτη ηλικία θα πάρεις κάτι που αναλογεί στο αναμενόμενο, στο, στο προσδόκιμο ζωής σου. Τώρα που οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωή από τους άντρες και βάσει αυτής της αρχής, της, της αναλογιστικής αρχής, οι γυναίκες πρέπει να ε, δουλέψουν τον ίδιο χρόνο με τους άντρες για να πάρουν τα ίδια, ωφελήμα, τα ίδια ωφελήματα ή να δουλέψουν παραπάνω όταν έχουν ε, φτάσει να είναι ηλικιωμένε, γιατί θα ζήσουν τελικά πολύ παραπάνω από τον αντίστοιχο άντρα, ενώ έχουν ίσα εισοδήματα από τη σύνταξη. Κάτι άλλο που έχει συμβεί με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της συντάξης είναι η άνοδος του ορίου συνταξιοδότησης και η ε, εξίσωση του ορίου αυτού μεταξύ άντρων και γυναικών. Αυτό είναι κάτι το θετικό ω προ τα ωφελήματα, τα συνταξιδοτικά δικαιώματα. Διότι οι γυναίκε μπορούν να καταβάλουν εισφορέ για περισσότερο καιρό, όμω αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι οι γυναίκε θα πρέπει να δουλέψουν περισσότερο χρόνο, οπότε όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την φροντίδα εγγονιών, ηλικιωμένων γονέων, δεν αντιστοιχούν, δεν αναλογούν σε κάτι. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν πολιτική που να ε, ενισχύει του άντρε και τι γυναίκε που απασχολούνται σε υπηρεσίε με φροντίδα, αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και αν δούμε το ποσοστό απασχόληση των μεγαλύτερων γυναικών σε σχέση με του πιο ηλικιωμένου άντρε, οι γυναίκε έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό απασχόληση, διότι συνήθω παίρνουν σύνταξη νωρίτερα προκειμένου να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα εγγόνια του ή να φροντίσουν του ηλικιωμένου γονεί του. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να εξισορροπήσουν τρόπον την αυτές τις, αρνητικές, ε, τις ενδεχόμενες αρνητικές ε, συνέπειες λόγω των πρόσφατων συνταξιδοτικών μεταρρυθμίσεων. Και αυτά έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τις ε, αναλογικές πιστώσεις σύνταξης. Κάποια κράτη δηλαδή κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας ή της γονικής άδειας προσφέρουν κάποια ωφελήματα ε, με βάση τη φροντίδα που προσφέρεται. Αυτά διαφέρουν πολύ μεταξύ των χωρών, αλλά θα ήταν σκόπιμο να έχουμε ανταλλαγή των πρακτικών και μια ε, καλή σύγκριση μεταξύ των χωρών για να δούμε πού ε, η διευθέτηση αυτών των απιστώσεων θα πάει καλύτερα για να μειώσει και να αμβλύνει τι ανισότητε μεταξύ των δύο φίλων ω προ τα συνταξιδοτικά ωφελήματα. Ένα πρόβλημα με αυτέ τι περιπτώσει που σχεδόν όλε οι χώρε το βλέπουν είναι ότι οι πιστώσει για τα παιδιά, για τη φροντίδα των παιδιών είναι πολύ χαμηλότερε. από ό,τι για του ηλικιωμένου. Να άλλο ένα τομέα, όπου ίσω κάτι θα μπορούσε να γίνει. Ε, κάτι ακόμα είναι η πιο περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στα ε, ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό. Οπότε και πάλι εδώ κάτι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιώσουμε την πρόσβαση των γυναικών σε αυτά τα συστήματα, τα ταμεία και ο, η διευθέτησή του, ο τρόπο που λειτουργούν να γίνει πιο φιλικό προ τι γυναίκε. Συνήθω τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία έχουν σεξιστ η προσέγγιση στα, στις τιμές τους, δεν προσφέρουν κάποια κάλυψη στην περίπτωση της φροντίδας, ούτε τα ανάλογα ωφελήματα μετά στη σύνταξη. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα στα ιδιωτικά συνταξιδετικά ταμεία να είναι πιο φιλικά προς τις γυναίκες από ό,τι είναι τώρα. Τέλος, ο τρίτος τομέας όπου έχουν ως τώρα υπάρξει αλλαγές έχουν υπάρξει σοβαρές έχει υπάρξει σοβαρή συνεισφορά στην κάλυψη του συνταξιδοτικού χάσματος είναι το τι γίνεται με τις επιβιώσεις συντα... συνταξιούχους, γυναίκες που αυτή τη στιγμή παίρνουν σύνταξη και τι σύνταξη λαμβάνουν. Εδώ έχουμε ένα τομέα που και πάλι μπορεί να χρειαστεί παρέμβαση. Είναι ένα θέμα σαφώ αμφιλεγόμενο, διότι από τη μια πρέπει να δώσουμε κίνητρα στι γυναίκε να παντρευτούν. προκειμένου σε μεγαλύτερη ηλικία να είναι σε θέση να έχουν το κατάλληλο δικαίωμα, το δικαίωμα μέλους οικογένειας, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί για τις γυναίκες που ε, είναι μόνες και δεν έχουν παντρευτεί. Είναι ένα κίνητρο δηλαδή που κάνει μια διάκριση μεταξύ των παντρεμένων και των ανήπαντρων. Οπότε, μια και το ποσοστό των ανήπαντρων αυξάνεται ε, σημαντικά, ιδίω μεταξύ των νέων, και αν θέλουμε να σκεφτούμε τους μελλοντικού συνταξιούχου, θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το τομέα, ε, μάλιστα διεξοδικώς. Υπάρχουν συνδεξιδικά ωφελήματα που δεν αφορούν μόνο τα, τις συντάξεις χειρίας, αλλά και αυτά από... Ε, από διαζύγια, από γυναίκες που συντηρούν μόνο στους μια οικογένεια ενώ χωρίσανε και ούτω καθεξής. Ε, εάν τώρα δούμε το χάσμα, το συνταξιδοτικό προς τα φύλλα, Ήδη το περιέγραψε η συγκητρία, όπως σας είπα. Πρώτη φορά εκτιμήθηκε το 2013 από ε, τον BPO και άλλους. Τώρα ε, υπάρχουν πολλές εκθέσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αυτή που σας παρουσιάζουμε εμείς αφορά προέρχεται μάλλον από την υπηρεσία ισότητας των φίλων της Γενικής Διεύθυνσης JAST, η οποία παρουσιάζει έκθεση για την ισότητα των φύλων ε, μια φορά το χρόνο. Καλό θα ήταν εδώ να πούμε ότι αυτό το χάσμα ε, μεταξύ των δύο φίλων στις συντάξεις καταγράφει τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών και το μέσο του εισόδημα βάσει της σύνταξης. Δηλαδή μιλάμε για συνταξιδοτικά δικαιώματα. Αυτή η εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι περίπου 40,2% κατά μέσο όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Εάν λάβουμε υπόψη όλους τους ηλικιωμένους, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν συνταξιδοτικά δικαιώματα, το συντεξιδοτικό χάσμα αυξάνεται πολύ περισσότερο. Πολλές γυναίκες δεν έχουν κανένα συντεξιδοτικό δικαίωμα, διότι δεν δούλεψαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους κατά βάση, όταν ήταν νεότερες. Όπω βλέπετε εδώ και ήδη υπόθηκε και προηγουμένω από την εισηγήτρια, το χάσμα αυτό βαθαίνει, μεγαλώνει όταν υπάρχει και το ανάλογο μισθολογικό νωρίτερα. Διότι το σύστημα των συντάξεων μπορεί να εντείνει διαφορές που ούτως ή άλλως υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Δηλαδή διαφορές μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, τι απολαβές και ούτω καθεξής. Εάν δούμε τις διαφορές μεταξύ των κρατών, κάτι άλλο που προκύπτει από το χάσμα μεταξύ των φίλων της συντάξεις, είναι ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις μεταξύ των χωρών. Από 3-4% στην Εστονία σε πάνω από 40% στην Κύπρο. Οι διαφορές είναι έντονες. Είναι βαθιές και πολλές φορές οι διαφορές στο συνταξιδοτικό αντικατοπτρίζουν και διαφορές επίπεδο κράτους ε, λόγω της εθνικής αγοράς εργασίας όπως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι μικρότερο από ό,τι στις πλούσιες δυτικές χώρες. Αυτό δείχνει διαφορές στο πόσο είναι διαδεδομένη η απασχόληση μερικού χρόνου μεταξύ των γυναικών. Υπάρχουν χώρε όπου είναι τόσο διαδεδομένη η εργασία μερική απασχόληση μεταξύ των γυναικών είναι τεράστιο μισθολογικό χάσμα. Η Εστονία έχει πολύ χαμηλό μισθολογικό χάσμα, ακόμη και αν μάλλον ε, χαμηλό χάσμα, ακόμη και αν έχουν τεράστιο μισθολογικό. Ε, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη το μισθολογικό του. Όμω το σημερινό του συνταξιδοτικό σύστημα για του συνταξιούχου όλου είναι αρκετά γενναιόδωρο ακόμη και για τι γυναίκε και με πολύ χαμηλά ε, χρόνια ε, εισφορών και πολύ χαμηλό εισόδημα. Έχουν ε, βασική ελάχιστη σύνταξη βάσει τη κατοικία του που είναι αρκετά γενναιόδωρο σε σχέση με όσα ισχύουν στα υπόλοιπα συνταξιδοτικά τώρα. Επίσης να πω κάτι που ξέχασα να πω προηγουμένως, ότι όταν μιλάμε για συνταξιδοτικό χάσμα είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ της κατάστασης που επικρατεί ε, σε όσους τώρα είναι συνταξιούχοι, στην τρίτη ηλικία, που επηρεάζονται από ισχύοντας τα προηγούμενα συνταξιδοτικά συστήματα και ενδεχομένως και από τις τωρινές εξελίξεις στα δικαιώματα, σε ωφελήματα βάσει των περικοπών στις κρατικές δαπάνες λόγου χάρη και να το δούμε σε διαστολή με την κατάσταση των μελλοντικών συνταξιούχων που θα επηρεαστεί ιδιαίτερο από τις μεταρρυθμίσεις των συνταξιδοτικών συστημάτων που σας ανέφερα προηγουμένως. Και αυτοί πάντως θα αλλάξουν μάλλον τη συμπεριφορά τους στην αγορά εργασίας βάσει αυτών των συνταξιδοτικών μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσουν την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία στο μέλλον, κατά πάσα πιθανότητα. Ιδάλω, θα έχουμε πολύ λιγότερα συνταξιωτικά ωφελήματα από ό,τι έχουν οι τωρινοί συνταξιούχοι. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Το πρόβλημα είναι ότι τις νεαρές γυναίκες ε, που θα είναι συνταξιούχοι στο μέλλον θα είναι πρόθυμες να δουλέψουν παραπάνω, να δουλέψουν σε ε, θέσεις ε, πλούρης απασχόλησης, αλλά το ερώτημα είναι αν θα είναι σε θέση να το κάνουν. Ε, σε κάποια κάτι μέλη δεν υπάρχουν καθόλου μέτρα για να τις υποστηρίξουν. Για να εργαστούν σε πλήρη απασχόληση, να εργαστούν για πιο πολύ καιρό, τουλάχιστον 40 χρόνια, για να καταβάλουν και τις εισφορές τους, Οπότε θα ε, ε, έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε αντί να περιοριστεί θα ενταθεί το συνταξιδοτικό χάσμα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, ένας άλλο σημαντικός δείκτης, όταν μιλάμε για, τα, ε, για τις διαφορές στο συνταξιδοτικό χάσμα, είναι η κάλυψη. Η κάλυψη σε κάποιες χώρες ε, ε, έχει το εξή πρόβλημα. Κάποιες γυναίκες δεν έχουν συντεξιωτικά δικαιώματα. Ιδίως στις χώρες όπου υπάρχει το λεγόμενο μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή έχει κανείς δικαίωμα σε σύνταξη μόνο αν έχει δουλέψει τουλάχιστον για ένα χι αριθμό ετών. Πολλές γυναίκες που δεν έχουν αυτό το ιστορικό αυτό τον αριθμό ετών που απαιτείται, δεν, υπά... δεν καλύπτονται καν από το συνταξιδοτικό σύστημα. Κάποιες χώρες όπως η Μάλτα, η Ιταλία, η Ισπανία, Κάποιε χώρε έχουν πραγματικά πολύ μεγάλες ε, διαφορές ε, σε αυτό το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Οι περισσότερες όμως ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τεράστια διαφορά ως προς την κάλυψη των συντάξεων. Δεν είναι τεράστια δηλαδή διαφορά μεταξύ ως προς αυτό στην κάλυψη ανδρών ή γυναικών ως προς το κατά πόσο θεμελιώνεται συνταξιωτικό δικαίωμα. Στις χώρες όπου η κάλυψη είναι πολύ διαφορετική υπάρχει ούτως ή άλλως ανισότητα των φύλων. Αν δούμε δηλαδή συνολικά τον, ε, το τι συμβαίνει στο επίπεδο των ε, ε, τις ηλικίες των 65 ε, λόγω χάρη στην Ιρλανδία, την Ισπανία μιλάμε για 52% συνολικά προ προς την ανισότητα των φύλων, 49% συνταξιούχοι και μη συνταξιούχοι μαζί. Υπάρχει πρόβλημα ούτως ή άλλως. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω για να κλείσω κιόλα είναι να σας πω ποια είναι τα βασικά αίτια του συνταξιδοτικού χάσματο μεταξύ των δύο φύλων. Είδαμε ήδη κάποια από αυτά. Διαφορέ ε, στην αγορά εργασία μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή διαφορά ε, στην απασχόληση, στα έτη απασχόληση, στο χρόνο απασχόληση, μερική απασχόληση πολύ σημαντική συνιστόσα, το κατά πόσον οι εισφορέ καταβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου και αυτά θα αρχίσουν να αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία και να επηρεάζουν τα συνταξιδοτικά δικαιώματα σε πιο προχωρημένη ηλικία. Πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Εάν λοιπόν οι γυναίκες δεν βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ως προς τους άντρες, ε, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Και ε, το χάσμα αυτό ε, των δύο φίλων μας προς τις συντάξεις θα αυξηθεί. Επίσης η οικογενειακή κατάσταση, η μητρότητα, τα, οι υποχρεώσεις φροντίδας είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες, διότι είναι ακριβώς τα βασικά αίτια που εξηγούν γιατί οι γυναίκες έχουν διαφορετική συμμετοχή και διαφορετικές συνθήκες ε, και θέσεις στην αγορά εργασίας. Εάν δούμε το, τις διαφορές των φύλων από τη σκοπιά των γυναικών με παιδιά ή για τις ύπανδρες γυναίκες, αυτή η διαφορά αυξάνεται πολύ περισσότερο από ό,τι στο μέσο όρο. Και μάλιστα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Όσο πιο πολλά παιδιά έχει καμία, κάποια γυναίκα, τόσο λιγότερο μπορεί να έχει θέση πλήρου απασχόληση και το αντίστροφο. Εκτό κι αν υπάρχουν ειδικέ διατάξει στην νομοθεσία που να το επιτρέπουν. Επίση, ε, μπορεί η συμπεριφορά των νέων γυναικών που απασχολούνται στην αγορά εργασία, να ε, επηρεάσει το τι θα γίνει στο μέλλον, δηλαδή η απασχόληση των γυναικών, η καταβολή φορών, η θεμελίωση συνταξιδοτικού δικαιώματος και σχετικοί κανόνες σε κάποιες χώρες, όλα αυτά Όλοι αυτοί οι παράγοντε στο σχεδιασμό των συνταξιδοτικών συστημάτων, εφόσον ληφθούν υπόψη, μπορούν να καλύψουν το χάσμα σε έναν βαθμό. Σε κάποιε χώρε που δεν λαμβάνονται υπόψη, που δεν υπάρχει καλή διευθέτηση, το χάσμα είναι πολύ πιο έντονο. Ποιε είναι οι επιπτώσεις ως προς τους κινδύνους να βρεθεί κανείς στα όρια της φτώχειας και την κάλυψη. Το ποσοστό φτώχειας για τους συνταξιούχους, όχι για τον συνολικό πληθυσμό, για τους ανθρώπους που έχουν συνταξιωτικό δικαίωμα. Υπό μία έννοια αυτές είναι οι γυναίκες που έχουν σύνταξη, που θα έπρεπε να είναι σε καλύτερη θέση από τις γυναίκες που δεν έχουν καν σύνταξη. Και πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων υπάρχει κίνδυνο να περάσει κανεί τα όρια τη φτώχεια και για συνταξιούχου. Όπω είπα προηγουμένω, οι γυναίκε συνήθω έχουν πρόσβαση στην ελάχιστη σύνταξη. Σε πολλέ χώρε οι ελάχιστε αυτέ συντάξει είναι χαμηλότερε του εισοδήματο που είναι χαμηλότερε του ορίου φτώχεια. Δηλαδή, έχουν σοβαρότατο κίνδυνο να περάσουν το όριο τη φτώχεια. Για να συνοψίσω, Κάναμε και μία μελέτη για το τι έχει γίνει στην Ευρώπη, σε κάποια κάτι μέλη, ως προς την καλλιέργεια μεγαλύτερης ισότητας για να καλύψουμε το συντεκδοτικό χάσμα, ιδίω με βάση το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα πολύ ε, σημαντικό εργαλείο οικονομικού συντονισμού ε, με κυκλικό χαρακτήρα και με συστάσεις αναχώρα. Στι συστάσεις αναχώρα 2012-2015 οι συντάξει αναφέρονταν στο 10% του συνόλου των κειμένων των αναχώρα συστάσεων. Ωστόσο, ουδέποτε ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε αυτές τις, αναχώρασει τις αναχώρασεις τάσεις ε, και στις αναφορές στις συντάξεις στο σκέλος της, των διαφορών των φύλων, των ανισοτήτων των φύλων. Πολύ λίγη προσοχή δόθηκε στην ανάγκη να στηριχθούν οι γυναίκες ως προς τα εισοδήματά τους στην απασχόληση και να καλυφθεί αυτό το συνταξιδοτικό χάσμα. Πολύ λοιπόν λίγη προσοχή για θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις και τις σχετικές πολιτικές. Επίσης, κανένας δείκτης για το συνταξιδοτικό χάσμα στη μακροοικονομική ε, μελέτη του scoreboard, του βαθμολογίου, αυτό είναι μια πρόταση που θα μπορούσε να προκύψει από το Κοινοβούλιο ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, να συμπεριληφθεί ένας δείκτης, όπως αυτός που έχουμε συζητήσει και που ήδη χρησιμοποιείται πολύ στο βαθμολόγιο για την μακροοικονομική εποπτεία διότι στον πίνακα βαθμολογίας οι δείκτες αυτοί καταλήγουν να είναι πολύ σημαντικοί. Όλη η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του πολιτικού συντονισμού και των ανασυχώρα συστάσεων ε, πρέπει να, να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις των δικτών. Επίσης, η πρόταση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στα συνταξιωτικά συστήματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου προκειμένου να σχεδιαστούν σωστά οι μεταρρυθμίσεις. Για να ολοκληρώσω και ως προς τις πολιτικές κατευθύνσεις, κατά πρώτον, ε, σαφώς υπάρχει ανάγκη πρώτα απ' όλα να ε, υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασία. Ιδάλω δεν θα έχουν καλέ συντάξει. Καθόλου με το ισχύον σύστημα. Ε, Επίση όμω πρέπει να αναθεωρήσουμε και να ξαναδούμε τον σχεδιασμό των συνταξιδοτικών συστημάτων προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονό ότι οι γυναίκε έχουν ευθύνε και υποχρεώσει φροντίδα. Πολλέ φορέ δεν μπορούν να έχουν ε, δουλειά πλήρου απασχόληση και για όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία που απαιτείται για να θεμελιώσουν δικαίωμα. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε το αν θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τις καθολικές βάσεις της κατοικίας ελάχιστες συντάξεις, τις επικουρικές συντάξεις για γυναίκες, ε, τη βελτίωση των κανόνων και των νόμων για αυτά τα συστήματα προκειμένου να είναι πιο φιλικά προς τις γυναίκες. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε τις πιστώσεις των συντάξεων φροντίδας όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άντρες για να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση και στερεότυπα όπως στην αγορά εργασίας. Επίσης είναι μια άλλη σημαντική πτυχή. Αυτά Αυτές οι ενδείξεις δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες, αφορούν τους πάντες. Διότι με την ε, αύξηση του προσδοκίμου δε ζωής, από ό,τι φαίνεται θα μένουμε στην αγορά εργασίας πολύ περισσότερο. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι θα μπορούν οι άνθρωποι να μένουν αδιαλείπτως στην αγορά εργασίας. Υπό μία έννοια μπορεί να χρειαστεί μια προσέγγιση που να έχει να λάβει υπόψη να μπορεί να λάβει υπόψη της και την πορεία της ζωής ως προς τις συντάξεις. Δηλαδή οι περισσότεροι κατά διαστήματα θα εργάζονται, θα εκπαιδεύονται, θα βγαίνουν εκτός αγοράς εργασίας γιατί έμειναν άνεργοι, γιατί υπήρξε κρίση. Οπότε τα συνταξιδοτικά συστήματα εάν θέλουμε να είναι βιώσιμα, εκτός από βιώσιμα να είναι και αποτελεσματικά, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στην πορεία ζωής τους μπορεί κα... Μπορεί οι εργαζόμενοι να βρεθούν και εκτό αγορά εργασία για κάποιο διάστημα. Τα συνταξιδικά λοιπόν πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη. Κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ε, μέτρα για να στηριχθούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και να στηρίξουμε τις υποχρεώσεις φροντίδας. Λόγου χάρη η παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξη γυναικών με τέτοιες υποχρεώσεις και ευθύνες. Επίσης να στηρίξουμε τελειώνω, την, ε, της προσοχή, τη στόχευση πρέπει να δώσουμε στην ε, σκοπιμότητα των συντάξεων και την κάλυψη των συνταξιδοτικών διαφορών. Λόγω χάρη υπόθηκε ήδη με περισσότερες ε, ε στατιστικές που να έχουν συμπηλήσει σωστά τα δεδομένα και ε, συμπεριλαμβάνοντας αυτούς τους δείκτες που ανέφερα στη δικασία του Ευρωπαϊκού Ξαμήνου και επίσης επιβλέποντας πάντοτε εκ των προτέρων εξάντε ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στα εκλογικά συστήματα υπό την προοπτική του, ε, των δύο φύλων. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίω το Ευρωκοινοβούλιο, για να καλλιεργήσουν αυτήν την ε, πολιτική κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαντοβίτση για αυτή την ε, τόσο διεξοδική παρουσίαση σε αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Οι σκιώδεις εισηγητές έχουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση της μελέτης, να ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα και την εισηγήτρια η οποία ε, δημιούργησε τι εξαιρετικές προϋποθέσεις. Πιστεύω πως υπάρχουν δύο ειδών αδικίες στην Ευρώπη. Η πρώτη αδικία είναι φορολογική, το πώς φορολογούμαστε. Η δεύτερη μεγάλη αδικία είναι ο τρόπος ε, με τον οποίο γίνονται οι συνταξιδοτικές εισφορές, που δεν έχει καμία σχέση με τις επιδόσεις, με το τι κάνουμε. στις συντάξεις όσοι δουλεύουν πολύ δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα έχουν και, μεγάλες, ε, και μεγάλη σύνταξη. Και πιστεύω πως αυτή είναι μεγάλη, ε, η μεγάλη ανισότητα. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν ε, έχουν γίνει λάθη, υπάρχουν ανισότητες, διότι διαφορετικά αν το δούμε σύμφωνα με ε, τα στοιχεία θα πούμε ότι οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερο, άρα καλώς έχουν και μικρότερη σύνταξη. Όμως, το τι συνεισφέρει μία γυναίκα δεν υπολογίζεται ε, στην ολότητά του. Υπολογίζεται μόνο η επαγγελματική σταδιοδρομία, οι επαγγελματικέ εισφορέ και όχι οι εισφορέ στη φροντίδα τη οικογένεια, στην ανατροφή παιδιών κτλ. Και εδώ πιστεύω πω υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Όταν μια γυναίκα δουλεύει εθελοντικά, όταν μια ε, γυναίκα εργάζεται ανατρέφοντας τα παιδιά της, ε, ούσαν νοικοκυρά, σιδερώνοντας ρούχα, μαγειρεύοντα. Όσο περισσότερο λοιπόν μια γυναίκα δουλεύει αμυστή, με αυτόν τον τρόπο τόσο μικρότερη θα είναι και η σύνταξη που θα πάρει, ε, τόσο λιγότερο αναγνωρίζεται ε, αργότερα στην ε, ζωή της. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε πως η, το σύστημα των συντάξεων δεν είναι δίκαιο και αυτό το χάσμα στις ε, αποδοχές υπάρχει εξαιτία αυτών των ανισοτήτων. Υπάρχει ακριβώς επειδή αυτή η συνεισφορά των γυναικών δεν αμείβεται. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να αλλάξει ε, ριζικά το σύστημα, χρειάζεται να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, να... έτσι ώστε να έρθει ισότητα έτσι ώστε να κλείσει αυτό το ε, συνταξιδοτικό χάσμα. Να αναγνωριστεί δηλαδή αυτή η άμυστη εργασία των γυναικών. Ο στόχος πρέπει να είναι οι γυναίκες σε κάθε σημείο της ε, ζωής τους να μπορούν να ζήσουν είτε με το εισόδημά τους είτε με τη σύνταξή τους. Και αυτή τη στιγμή απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Το θέμα αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και πιστεύω πως ε, δεν υπάρχει μία εύκολη απάντηση και η συγγήτρια κιόλα ε, το ανέφερε, ήταν σαφέστατη. Υπάρχουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας, υπάρχουν διακρίσεις στην έμισθη και άμισθη εργασία. Το θέμα λοιπόν είναι πώς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να διορθωθεί αυτή η ανισότητα. Όσο στηρίζεται αυτή η ανισότητα, όσο στηρίζεται δηλαδή από τις πολιτικές των κρατών μελών το να μένει ένας γονιός στο σπίτι, όσο στηρίζεται από το φορολογικό σύστημα. Και να σας πω ότι στη Γερμανία το φορολογικό σύστημα υποστηρίζει ε, το να δουλεύει ένας μόνο από τους δύο γονείς και ο άλλος να κάθεται στο σπίτι. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η στήριξη από το κράτος αυτού του τρόπου ζωής δεν θα αλλάξει τίποτα. Και στη Γερμανία είναι πολύ έντονη αυτή η προτίμηση. Και είναι εξάλλου μια χώρα στην οποία παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ε, συνταξιδοτικές διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα σύνταξης ε, χειρίες, να υπάρχει δυνατότητα διαφόρων επιδομάτων ανατροφής παιδιών. Όμως αυτά ε, είναι μόνο βραχυπρόθεσμες ε, μεταβατικές λύσεις. Μακροπρόθεσμα χρειάζεται θεμελιώδης αλλαγή του συστήματος έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνεισφορές των γυναικών. Και τέλος να πω ότι ο καταμερισμός της ε, εργασίας δεν πρέπει να γίνεται πάντα εις βάρος των γυναικών. Αυτά λοιπόν ως προς τις δύο μεγάλες ανισότητες, φορολογική, συνταξιοδοτική, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές συνεισφορές των πολιτών. Και αυτό πρέπει απαραίτητος να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή συζητούμε για, για την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ανισότητας των συντάξεων. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε και το εξής, ότι οι ανισότητες δεν προκύπτουν από μόνες τους και ξαφνικά. Πάντοτε οι γυναίκες ε, για την ίδια δουλειά πληρώνονταν λιγότερο από τους άντρες. Ένας από τους κυριότερους λόγους για αυτό το ε, μισθολογικό χάσμα είναι το γεγονός όμως και ότι οι γυναίκες γίνονται μητέρες. Και αυτό τις φέρνει σε μειονεκτική θέση. Τις αναγκάζει να μείνουν στο σπίτι, να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους, να εργάζονται με μερική απασχόληση ή να εγκαταλείπουν εντελώς με το δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο παιδί τον επαγγελματικό στίβο και να αλλάξουν επάγγελμα, δηλαδή από επαγγελματίε να γίνουν μητέρες. Αυτό λοιπόν ε, θα το έλεγα καλύτερα οικογενειακό χάσμα, χάσμα οικογένειας, όχι χάσμα μισθολογικό θεωρούμε πως ε, το να είσαι γονιός πρέπει να αναγνωρίζεται ως επάγγελμα. Διότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα ήταν και η δαμόκλειο πάθη τα τελευταία χρόνια σε αυτό το μισθολογικό χάσμα. Πιστεύω πως λάθος προσανατολιζόμαστε στο ε, ποιος πρέπει να φροντίζει περισσότερα τα παιδιά, ποιος λαμβάνει περισσότερα, ε, περισσότερη αμοιβή. Αλλά πρέπει να δούμε ότι η διαφορά, το χάσμα, εστιάζεται ανάμεσα σε άτομα που έχουν παιδιά και σε άτομα που δεν έχουν παιδιά. Και αυτό δεν είδα να αναφέρεται πουθενά, ούτε στη μελέτη το είδα να αναφέρεται. ότι οι μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα σε ε, γυναίκες με παιδιά. Χρειάζεται λοιπόν μια διαφορετική αντιμετώπιση, μια διαφορετική θεώρηση του προβλήματος, ε, το να θεωρούνται οι γονείς επαγγελματίες, εργαζόμενοι. και θα πρέπει να αναλογιστούμε το ότι ίσως θα έπρεπε να αμείβονται οι γονείς, οι μητέρες ή οι πατέρες ακριβώς για το γεγονός ότι εργάζονται στην ανατροφή των παιδιών τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν είναι εδώ κυρία Μπίρντερ, οπότε Θα αφήσω για το ρόλο του Προεδρεύοντα και θα μιλήσω ως και ο για να εκφράσω και εγώ τις παρατηρήσεις για αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Για το θέμα λοιπόν αυτό μας φαίνεται καθοριστικής σημασίας να δοθεί έμφαση αυτή η διπλή, για να μην πω πολλαπλή, διάκριση βάρος των γυναικών να βρεθεί και να εκφραστεί ανάγλυφα για να δούμε τα γενεσφυρουργά αίτια ε, του συνταξιδοτικού χάσματο λόγω τη διάσταση των διαφορετικών φύλων. Και ω προ την απασχόληση. Οι γυναίκε, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκε, βρίσκονται να είναι θύμα διακριτική μεταχείριση επειδή είναι μητέρε, επειδή θέλουν να γίνουν μητέρε, και σε αυτά προστίθεται η διακριτική μεταχείριση σε επίπεδο μισθού, απολαβών και αποσχόλησης και πρόσβασης στην αγορά. Οι γυναίκες εδώ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και ε, ο δείκτης διακριτικής μεταχείρισης είναι πολύ ε, σημαντικότερος από ό,τι στους άντρες, πολύ πιο μεγάλος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κοινωνικό στίγμα, κοινωνικό στιγματισμό, ε, κοινωνική διακριτική μεταχείριση στι εργασιακέ σχέσει και βεβαίω αυτό ξύνεται ε, λόγω τη διάσταση των φύλων. Το γεγονό ότι κάποιος, μια γυναίκα μάλλον, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα, έχει διπλές, ε, διπλά στοιχεία εις βάρος της. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, δούμε βάσει των πορισμάτων και μιας μελέτης και της συγκεκριμένη μελέτης ε, αυτό που προκύπτει ότι οι γυναίκες για να έχουν το ίδιο επίπεδο σύνταξη με βάση τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να δουλέψουν περισσότερα χρόνια από τους άντρες για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι πραγματικά σχεδόν ε, προσβλητικό και είναι και παράλογο, διότι από όλη αυτή την προσπάθεια ε, άμβλυνσης της διακριτικής συμπεριφοράς, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου, ε, ουσιαστικά του αφαιρεί όλη την ε, λογική του. Ε, εάν έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός ε, συνταξιοδότησης σε κάποιες χώρες, όπως τη δική μου λοιπόν τη χώρα, επειδή είμαι Πορτογάλος, στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή το χρήμα που καταβάλουμε για τις συντάξεις δεν παραμένει σε κάποιο ταμείο. Δεν μας περιμένει για την ε, κατοπινή ζωή μας, για τη μεγάλη ηλικία. Αυτή τη στιγμή σφαίρουμε για τους σημερινούς συνταξιούχους άντρες και γυναίκες. Οπότε η μεταρρύθμιση που θα γίνει και θα καλύψει τη δική μας σύνταξη σε μερικά χρόνια σημαίνει ότι θα βρεθούμε σε διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης και θα ισχύουν όλα αυτά για όσους δουλέψουν τώρα. Οπότε δεν μπορούμε να ξεχνάμε τον αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά, ε, που έχουν σε όλα αυτά οι πολιτικές λιτότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τώρα ε, ε, επικρατήσει οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν πρόσφατα, η ιδιωτικοποίηση των συνταξιδοτικών ταμείων, ενώ θα ήταν δυνατόν να καλυφθούν οι μισθολογικές αποκλήσεις εάν υπήρχε ένα σύστημα ε, εισφορών για τις συντάξεις που να είναι προοδευτικό. Όποιος ε, κερδίζει περισσότερα να πληρώνει περισσότερα και όποιος κερδίζει λιγότερα να καταβάλει λιγότερα. Αυτό για να ανακεφαλαιώσω και να πω ότι θα έπρεπε να ξεπεράσουμε αυτές τις ανισότητες από την εξέταση του όλου θέματος και από τις ιδεολογίες τις οποίες πιστεύουμε ότι τις ανέφερε και κάποιος προηγουμένως και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την επισφαλή εργασία. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις ως αποτελεσματικό μηχανισμό για να αμβλυνθούν αυτές οι ανισότητες, είτε είναι ακρεφνώς κοινωνικές είτε είναι ανισότητες φύλου. Πρέπει να προωθήσουμε την ισότητα στους μισθούς, δηλαδή την αρχή ίσως μισθός για ίση εργασία. Θα πρέπει να σχεδιαστούν εργαλεία για την άδεια ε, πατρότητας, μητρότητας, ε, τη γονική, ε, που να είναι τελείως αμοιβόμενες και να αποφεύγουν τις διακριτικές μεταχειρήσεις, τις διακριτικές μεταχειρήσεις που τόσο συχνά βλέπουμε να συμβαίνουν σε περίοδο ε, μητρότητα για τι γυναίκε. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκατέλειψε την οδηγία για την άδεια μητρότητα. Πρέπει να την ξαναδεί και να την ξαναπροωθήσει. Επίση, ο κοινωνικό ρόλο του κράτου πρέπει να ενισχυθεί, ιδίω ό,τι αφορά την ε, κρατική παροχή υπηρεσιών και εγκαταστάσεων που να διευκολύνουν ε, την ε, οργάνωση του οικογενειακού βίου και να αποφεύγουμε αποφεύγουμε τι ενσώτες και την διακριτική μεταχείριση που εδώ αναφέρθηκαν. Οι γυναίκες πολλέ φορέ αναγκάζονται να φροντίσουν παιδιά και συγγενεί. Αυτό ήταν το τέλο τη παρεμβασή μου. Θα δώσω τώρα το λόγο, όπως προβλέπετε, στην εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης, Τάνια Γκονζάλεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ε, πρόσκληση στην σημερινή συνεδρίαση ως εισηγήτρια της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η οικονομική ανισότητα ανδρών και γυναικών απορρέει από διάφορους παράγοντες, ο πιο σημαντικός ε, εκ των οποίων είναι το χάσμα το συνταξιωτικό. Σημερινή κατάσταση που ναι μεν ποικίλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος αλλά έχει τον μέσον όρο αυτό απόκληση 38%. Σε σχέση με την πρόσβαση σε υπηρεσίες και ισότητα ανδρών και γυναικών 34 και 23 άρθρα της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπως και σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμήσει τις διακρίσεις και την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα λοιπόν, παρότι η δομή και ο σχεδιασμός των συνταξιωτικών συστημάτων είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτούς τους στόχους εκπεφρασμένα και επομένως θα πρέπει να έχει και ένα επαρκές επίπεδο προστασίας κοινωνικής, όπως λέει και το άρθρο 51 της δίκης. Υπό αυτή, θα πρέπει να συμπληρώνει και να επικουρεί τη δράση των κρατών μελών, μια και εγγράφονται στα θεμελιώδη δικαιώματα και στη χάρτα. Παρά τα αυτά, η γραμμή που ακολουθείται τελευταία χρόνια αποκλίνει από το στόχο αυτό. Οι μεταρρυθμίσεις των εθνικών συστημάτων συνταξιοδότησης σχετικά με την... Ε, είναι, μάλιστα και η στροφή προς την ενίσχυση των ιδιωτικών ταμείων όπως έχουμε δει και από διάφορες, διάφορα σχόλια που έχουν υποβληθεί είναι μια, κατά την άποψή μας, ε, μια λανθασμένη ερμηνεία βιωσιμότητος. Έχουμε και τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επί των συνταξιών, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο επί των γυναικών. Και κάθε μεταρρύθμιση που γίνεται και που επιφέρει μεγαλύτερη επισφάλεια σύμφωνα με τα ίδια αυτά απορίσματα, καταλήγει σε νεότερη αρνητική επίδραση, αν θέλετε, για το επίπεδο των συνταξιωτικών ασόδων των γυναικών. Ίσως η κυρία Λοντοβιτσί μπορεί να μας το πει. Ίσως σύμφωνα με το όριο συνταξιοδότησης θα επέτρεπε μεγαλύτερα, περισσότερα χρόνια εργασίας για τις γυναίκες. Από την άλλη όμως, σύμφωνα με την τελευταία τουλάχιστον ισπανική μεταρρύθμιση, σήμερα προκειμένου να έχει κανείς πρόσβαση στην μέγιστη σύνταξη θα ήταν απαραίτητο να εργάζεται κανείς από τα 26,5 έτη ηλικίας χωρίς καμία διακοπή, το οποίο είναι απολύτως αδύνατον υπό τις σημερινές ε, συνθήκες εργασίας και ζωής. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο μειώνονται οι πιθανότητες και δυνατότητες να έχει μια γυναίκα πρόσβαση σε υψηλά επίπεδα συνταξιοδότησης. Έχουμε και τα θέματα της ε, διάκρισης, ε, των διακρίσεων κατά των γυναικών στο χώρο εργασίας, το οποίο συσχετίζεται όπως ε, είπαν και οι ομιλήτριες με το φαινόμενο της, ε, του χάσματος ε, του συνταξιωτικού. Έχουμε και τις διακρίσεις οριζόντιες και κατακόρυφες στον χώρο εργασίας, διάφορες άλλες διακρίσεις έμμεσες όπως λέγονται, οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί στις συλλογικές διαπραγματεύσεις γιατί όταν έχουμε διπλό άχθος, διπλή επιβάρυνση για τις γυναίκες πέρα δηλαδή από τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους για τη φροντίδα των ε, ε, πιο ηλικιωμένων μελών της οικογένειας και άλλες συμπληρωματικά καθήκοντα ε, συνεισφέρουν στα φαινόμενα μερικής απασχόλησης των γυναικών και όλα αυτά μαζί αθροισμένα οδηγούν αν θέλετε σε μεγαλύτερη αντετεκοποίηση του, των γυναικών εντός του πληθυσμού που είναι εκτεθειμένος ε, στην οικονομική επισφάλεια. Ε, και γι' αυτό θα θέλαμε να υποβάλουμε μια σειρά από προτάσεις μεταξύ των οποίων τις εξής να διευκολυνθεί, να, μάλλον να, ισχυθεί το, να ενισχυθούν τα δημόσια συστήματα εισφορών ή να εγκατασταθεί ένα σύστημα βαθμιαίων σταδιακών εισφορών αντί να διορθώνονται προς, προς τα κάτω τα επιδόματα και οι συντάξεις να υπάρχει καλύτερος σχετισμός ε, ετών εργασίας ανάλογα με τα παιδιά που έχει κάθε γυναίκα ή κάθε οικογένεια και επίσης τα εξαρτημένα άτομα που έχουν μερική απασχόληση να, ε, μετρά, το, να μετρούν τα ίδια εργασίες τους ως πλήρης εργασία, πλήρης απασχόληση. Αθρισμένα δηλαδή. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη συγχρηματοδότηση προκειμένου να ε, ενισχύσουμε τα μη ε, τα συστήματα, τα συνταξιοδοτικά που δεν βασίζονται στις φορές, μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Κοσλόφσκα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ε, ικανοποιημένοι που μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Για το συνταξιδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, ευχαριστώ την κυρία Λεγκρίπ για την τόσο καλή έναρξη όλης αυτής της συζήτησης και συγχαρητήρια και στην κυρία Λοντοβίτση για την εξαιρετική της ε, παρουσίαση εδώ. Πραγματικά ε, μας ε, φώτισε όλες τις λεπτομέρειες αυτού του τόσο πολύπλοκου ζητήματος. Εδώ λοιπόν ήθελα να θέσω ρωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ζήτησα μάλιστα το συνταξιδοτικό χάσμα να συμπεριληφθεί ως δείκτη στη δίκαση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να καλύψει και να αντικαταστήσει το μισθολογικό χάσμα, το σχετικό δίκτυο γιατί αφορά ολόκληρη την επαγγελματική σταδιοδρομία μιας γυναίκας ε, και δείχνει πόσο ασταθείς μπορεί να είναι οι δείκτες ε, στην προσπάθεια να αντικατοπτρίσουν την πραγματικότητα. Ε, το μισθολογικό χάσμα είναι ένας ε, πρώτος δείκτης, όμως η πραγματικότητα, πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται πολύ καλύτερα από τον δείκτη για τις διαφορές και τις ανισότητες στις συντάξεις. Ένας από τους λόγους των διαφορών στις συντάξεις ανδρών και γυναικών είναι η διαφορετική συμμετοχή στην αγορά εργασία. Οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερα από τους ε, άντρες. Επίσης, συχνά ε, κάνουν διακοπές, γιατί διαλύματα δηλαδή για να φροντίσουν τα παιδιά τους ή άλλου συγγενείς, άλλα μέλη της οικογένειας, ένας άρρωστος συγγενής, ένας γονιός. Οπότε, ούτως ή άλλως έχουν περάσει από διαφορετικά μονοπάτια εκπαίδευσης. Υπάρχει επίσης η αλλου συγγενεις αλλα μελη της οικογενειας ενας αρρωτος συγγενης ενας γονιος οποτε ουτως η αλλως εχουν περασει απο διαφορετικα μονοπατια εκπαιδευσης υπαρχει επισης η ταση οι γυναίκες να απασχολούνται σε θέσεις που αμείβονται χειρότερα και υπάρχει και η μισθολογική διαφορά από πάνω. Ένας μόνο από τους παράγοντες, αλλά είναι τόσες πολλές οι διαφορές. Ε, τόσες πολλές διαφορετικές συμπεριφορές ε, των γυναικών στην αγορά απασχόληση και ο τρόπος που απασχολούνται, που καταλήγουμε και σε άλλο χάσμα. Οι γυναίκες πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους ή τους ηλικιωμένους. Αυτή είναι η βασική λόγη των διαφορών και μπορούν να ληφθούν υπόψη. Μια από τι βασικέ λύσει είναι να δοθεί στις γυναίκες η δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτες στην αγορά εργασία. Η πρόταση τη Επιτρόπου Γιούροβα για περισσότερη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασία προκειμένου να βρουν τη σωστή ισορροπία επαγγελματικού και αγνοκοβίου είναι ήδη μια αρχή. Α μην ε, ε, πειράξουμε όμω τα συστήματα. Α επιτρέψουμε στις γυναίκε να ε, έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι απλώς ότι οι γυναίκες παίρνουν χαμηλότερη σύνταξη, είναι ότι κάποιος τις πληρώνει και λιγότερο για την ίδια εργασία που προσφέρει ένας άντρας. Πρέπει λοιπόν εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να πείσουμε τις γυναίκες να θεμελιώσουν συνταξιδοτικό δικαίωμα, να έχουν συντάξεις. Ε, Υπάρχει χάσμα σε πολλά επίπεδα. Να τους προσφέρουμε δημόσιες υπηρεσίες όπως ε, επέκου σταθμούς, ε, οίκου ευγυρίας, ε, υπηρεσίες φροντίδας που να τις επιτρέψουν να απασχολούνται όπως πρέπει. Επίσης, υπάρχει μεγάλη διαφορά λόγω και της μη αμοιβόμενης οικιακής εργασίας. Δεν λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουμε γι' αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε μια, ένα κατάλληλο σημείο ισορροπίας και να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, οι γυναίκες πολλές φορές δουλεύουν 10 ώρες παραπάνω την εβδομάδα από τους άντρες. Πρέπει και αυτό κάπως να το εξισορροπήσουμε και να λαμβάνεται υπόψη στην εξίσωση. Δεν γίνεται να μην πληρώνονται για αυτή τη δουλειά ή κάπως να μην αμείβονται. Επίση, η αμοιβόμενη φροντίδα των παιδιών είναι κάτι διαφορετικό. Εάν μιλάμε για οικογένειε με 5 και 6 παιδιά, ε ναι, σε μια τέτοια περίπτωση οι γυναίκες δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Μπορεί να χρειαστεί να τις πληρώνουμε για τη φροντίδα των παιδιών. E, για να ολοκληρώσω, για την αντιστάθμιση της φροντίδας των παιδιών και την καταβολή ε, εισφορών από τον κρατικό προπολογισμό. Αυτά σε έναν βαθμό γίνονται. Υπάρχουν ε, γονικές άδειε σε πολλές χώρες, όμως α μην μιλούμε για ε, παράταση των περιόδων αυτών, ε, τις αμοιβόμενες άδειες, διότι αυτό ε, βγάζει τις γυναίκες εκτός αγοράς εργασίας. Και είναι ένα από τα γενεσιουργά αίτια της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, οι γυναίκες στην ουσία δεν φτάνουν ποτέ στην ίση εργασία πλήρους απασχόλησης. Ευχαριστούμε κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λεγκρίπ για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντική και μας αφορά άμεσα. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Πέρα από τις προτάσεις σας, που αποτέλεσαν και αφορμή για συζήτηση σήμερα, έχουμε να εξετάσουμε επίσης και την ελάχιστη σύνταξη. Ελάχιστη δημόσια σύνταξη. Γνωρίζω πως ε, δεν είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου, είναι αρμοδιότητα εθνική το θέμα αυτό. Όμως ε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάποιες συστάσεις. Εγώ προσωπικά μελέτησα πάρα πολύ το θέμα των ελάχιστων συντάξεων και είδα ότι δεν υπάρχουν ίδιες ρυθμίσεις σε όλα τα κρατημέλη. Σε ορισμένα υπάρχουν τεράστιες διαφορές λόγω των διαφορετικών συνθήκων, των διαφορετικών εισφορών. Και λόγω των διαφορών αυτών πολλές γυναίκες βρίσκονται ε, στα όρια της φτώχειας. Στην Κροατία πολλές γυναίκες λαμβάνουν συντάξεις ε, που τις κάνουν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Με τα βίας επιβιώνουν δηλαδή. Και σε πολλές ανατολικοευρωπαϊκές χώρες η κατάσταση είναι παρόμοια. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της εκθεσή σας λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συμπεριλάβετε όλες τις ε, πτυχές και την ελάχιστη σύνταξη, η οποία δεν θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας, έτσι όπως αυτά ορίζονται από την Eurostat. Επίσης, οι γυναίκες της υπαίθρου δεν λαμβάνουν σύνταξη. Ακόμα και όταν εργάζονταν στην οικογενειακή τους ε, επιχείρηση, στην ε, οικογενειακή τους γεωργική εκμετάλλευση, δεν λαμβάνουν σύνταξη. και δεν βρίσκονται λοιπόν εντός του συνταξιδοτικού συστήματος. Ως κατά συνέπεια δεν λαμβάνουν σύνταξη και αυτή είναι μία ακόμα ομάδα την οποία πρέπει να λάβετε υπόψη θεωρώ και ε, συγχαρητήρια άλλη μια φορά. Ε, να δώσω και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Νταγκουάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Να υπογραμμίσω απλώς ότι οι αναλύσεις ε, της κυρίας Σαμέκ ε, συμπίπτουν απολύτως με τις δικές μας αναλύσεις, με τις αναλύσεις της Κομισιόν. Αποτυπώνονται πράγματι μερικώς αυτές οι αποκλήσεις, είτε οι μισθολογικές, είτε του χρόνου εργασίας, είτε της διάρκειας της σταδιοδρομίας, αλλά τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα μπορούσαν είτε να διορθώσουν είτε και να εντείνουν δυστυχώς αυτές τις αποκλήσεις. Επομένως κάθε πρόταση και ιδέα σχετικά με την ε, αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού θα πρέπει να εγγραφεί και στην ε, γενικότερη προσπάθεια την ευρωπαϊκή σχετικά με το εισόδημα των ηλικιωμένων αλλά και εντός του πλαισίου της πολιτικής αντιμετώπισης των ανισοτήτων των μισθολογικών στην εργασία, στην ίση μεταχείριση ή στην απασχόληση και την εργασία. Έχουμε την οδηγία σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις σχετικές δηλαδή ή στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα, που διέπει και τις συντάξεις, όπως και την πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ε, πρόνοιας. Το θέμα της μισθολογικής απόκλησης είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν και στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ε, κοινωνικής ε, συνεργασίας και ισότητας μεταξύ των φύλων που είναι η προτεραιότητα υπαριθμών 2 εκεί. Εξού και παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εργασίες σας και την γνωμοδότηση που θα υποβληθεί. Να δώσω και το λόγο στο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ να προσθέσω και εγώ δύο λόγια από τη Μονάδα Κοινωνικής Προστασίας της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ να πω απλώς ότι υποστηρίζουμε απολύτως την ανάλυση αυτή όπως είπε και η Λουσή και συμφωνούμε με την ανάλυση σας Υπάρχει όμως ένα πρόσθετο στοιχείο που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ίσως ε, να ανησυχούμε περισσότερο για τα επίπεδα έμβιας παρότι τις αποκλίσεις αυτές. Διότι οι γυναίκες όχι μόνο έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο από τους άντρες, αλλά ζουν και για περισσότερα χρόνια με ασθένειες και αναπηρία. Και εδώ μιλούμε για φροντίδες υγείας στα πλαίσια της οποίας η χαμηλότερη σύνταξη μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Ο τρόπος που χρηματοδοτούνται αυτά είναι τελείως διαφορετικό στα κράτη-μέλη. Η διάρκεια λοιπόν της ε, φροντίδας υγείας που λαμβάνει ο κάθε άνθρωπος έχει άμεσο αντίκτυπο επί του υπολογισμού αυτού Κοιτούμε λοιπόν και την ε, μυθολογική απόκληση υπό την σκοπιά αυτή. Δεν έχουμε εργαλεία σχετικά ε, με, τον υπολογισμό των πιθανοτήτων ε, αυξητικής ή μειωτικής τάσης του φαινομένου, αλλά μπορώ να σας ε, εγγυηθώ ότι όταν θα έχουμε και την έκθεση επί των συνταξιδοτικών θα εστιαστούμε στο χάσμα αυτό παρακολουθώντας με μεγάλο ενδιαφέρον και τις δικές σας εργασίες. Αυτά και από πλευράς μου ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Ο χόρδη καθυστέρησε η πτήση του και έφτασε μόλις τώρα. Θα έλεγα λοιπόν αυτό το σημείο να το αφήσουμε για την αυριανή συνεδρίαση για να το αφαιρέσουμε τον απαραίτητο χρόνο και αν είναι για τα δύο λεπτά που μένουν να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Λεγκρίπ για τις τελικές της παρατηρήσεις. Ε, για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Τώρα, και προς την κυρία Λοντοβίση, Λοντοβίτση μάλλον, και προς τους υπόλοιπους συναδέλφους, αν έχει κάποιος συνάδελφος να θέσει ερωτήσεις, ας κάνουμε τα υπόλοιπα γραπτός και ας ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση με την παρέμβαση της εισηγήτης. Παρακαλώ. Oui, merci, ευχαριστώ, Πρόεδρε δεν θα τολμούσα να πω ότι κλείνω ένα τόσο σημαντικό θέμα συζήτησης. Πάντως όλες οι συνεισφορές έδειξαν την περιπλοκότητα, τη δυσκολία του αντικειμένου που έχει αντίκτυπο επί διαφόρων επιπέδων πολιτικής ε, και έχει και διακυβεύματα πολύ σημαντικά δεδομένων και των τάσεων γύρανσης του πληθυσμού γενικά των δημογραφικών τάσεων. Ε, επομένως, ε, πράγματι, η μελέτη δίδει πολύ ενδιαφέρουσα τροφή προσκέψη. Θα πρέπει να μείνουμε βεβαίως στις αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής και της Επιτροπής μας. Άκουσα τις διάφορες απόψεις και συνεισφορές των σκιωδών, τους οποίους και ευχαριστώ θερμός όπως και των υπολείπων συνομιλητών που έδωσαν εκ των διαφορών πολιτικών ομάδων διάφορες απόψεις. Εγώ θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να ενσωματώσω όλες αυτές τις απόψεις σχετικά με ένα θέμα το οποίο ίσως μέχρι στιγμής να μην ήταν το αντικείμενο της μέγιστης δυνατής προσοχής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιλαμβανόμαστε την, τον πλούτο των εισφορών και της δουλειάς που έχει γίνει επί του θέματος αυτού. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε από κοινού αυτή τη δουλειά, ώστε να σχηματίσουμε, να διαμορφώσουμε με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο το έγγραφο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση δείχνει ότι φαίνεται έντονε οι συζητήσει μα στο μέλλον, παθιασμένε, με όλε αυτέ τι παρεμβάσει που ακούσαμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε συμβαστικέ λύσει. Θα έλεγα να κηρύξουμε τη λήξη τη σημερινή συνεδρίαση, να ευχαριστήσω του συμμετέχοντε. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά του και του διερμηνείς και για την επόμενη που είχαν. Να μα δώσουν λίγα λεπτά παραπάνω για αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ.